ψωμί θα γίνει αύριο. Συνεχίζουμε με τη συζήτησή μας. Ένα λεπτό διακόπτουμε. Witam pana Θα ήθελα να ελέγξουμε κατά πόσο όλοι είναι παρόντες. Έχουμε τον νέο επίτροπο, τον εισηγητή, άρα μπορούμε να... την εισηγήτρια, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχουμε την έκθεση της Ντατσάν Οκτάβια Σάρμπου για τα βιοκτώνα και μία δήλωση της Επιτροπής για μία νέα πρόταση για την αναθεώρηση ως προς τη διάθεση βιοκτόνων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Σάρμπου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής είναι μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για την παράταση των βιοκτώνων προϊόντων μέχρι το 2014. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται και στην ψηφοφορία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφους που ε, συνεργάστηκαν για την μεταβατική αυτή περίοδο μεταξύ τριών θεσμικών όργανων. Τα βιοκτώνα προϊόντα λοιπόν θα πρέπει να μπουν στην αγορά νόμιμα και η οδηγία αυτή θα πρέπει να περάσει σε πρώτη ανάγνωση για να μην ξεπεράσουμε τα 10 έτη για την ε, ε, επανεξέταση των βιοκτώνων και την απόρσυρσή τους από την αγορά μέχρι, από το 2010. Η παράταση της προθεσμίας διασφαλίζει στα κράτη-μέλη τον κατάλληλο χρόνο αποτίμηση των προϊόντων μέχρι το 2014 όταν θα τεθεί σε εφαρμογή αναθεωρημένη οδηγία. Ένα άλλο που προτείνω είναι ο περιορισμός σε δύο έτη της δυνατότητας για περαιτέρω παράταση για τους εναπομένοντες ε, φακέλους, να μην έχουμε άλλη επιτροπολογία πέρα από αυτήν, έτσι ώστε να μην καθυστερήσει επαόριστον η όλη διεργασία. Αυτό είναι αναγκαίο στην περίπτωση που η οδηγία αυτή δεν θα αναθεωρηθεί μέχρι το 2014. Τα στοιχεία που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων αφορούν την τακτική του free riding χρήσης προϊόντων, δηλαδή άλλων εταιριών που καταγράφονται σε ένα άλλο κράτος μέλος, έτσι ώστε να υπάρχει παράταση χρήσης βιοκτώνων και οι τροπολογίες υπάρχουν και στο τελικό σχέδιο που θα ψηφιστεί αύριο στην Ολομέλεια. Μετά από την ψήφο της Ολομέλειας θα έχουμε την υποστήριξη του Συμβουλίου για να έχουμε ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σταύρος Δήμας έχει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής. Συγκήτρια κυρία Ζάμπρου για την επιμέλειά της και τη προσπάθειά τη προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση τροποποίησης οδηγίας 98/8 για τη διάθεση βιοκτώνων στην αγορά. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να αποδεχθεί τη συμβιβαστική δέσμη και ιδίω το σημείο που αφορούν την ανάγκη της παράτασης μεταβατικής περίοδου κατά τέσσερα αντί για τρία έτη, καθώς και τον περιορισμό κάθε περαιτέρω ε, παράτασης σε δύο έτη και έτσι να διευκολύνουμε ε, το πρόγραμμα της αξιολόγησης. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Άρχεται λοιπόν η συζήτηση. Προχωρούμε πολύ γρήγορα και δίνω στον Κρίστο Κράς την, ε, το, το λόγο. Δύο λεπτά από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Δήμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τόσο υψηλό επίπεδο υγείας και υγιεινής. Και βεβαίως αυτό συνεισφέρει η χρήση διοκτώνων ως ε, ε, ουσίες που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση καθώς σκοτώνουν τους φορείς ε, επικίνδυνων ασθενειών. Βεβαίως είναι απολύτως απαραίτητες αυτές οι ουσίες. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να επανεξεταστούν όλες. Λέτε πως χρειάζεται χρόνο και πως η εξέταση χρειάζεται περισσότερο χρόνο από όσο αρχικά έχει σχεδιαστεί. Ο κίνδυνος να χαθούν σημαντικές ουσίες γιατί δεν έχετε τελειώσει με την καταγραφή δεν είναι δυνατό να γίνανε. Εκτός γι' αυτό χαιρετίζω το ότι η Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν συμφώνησαν στην πρώτη ανάγνωση σε μια γρήγορη παράταση των προθεσμιών σχετικής ε, Οδηγία και μπορούμε να συμφωνήσουμε νομίζω στο 2014. Γιατί όμως έρχεται τόσο αργά αυτή η πρόταση. Γιατί βεβαίως ο κίνδυνος αυτός ήταν ορατός εδώ και καιρό. Και τελικά αναγκαστήκαμε να κάνουμε διαπραγματεύσει υπό την πίωση χρόνου. Υπήρχε εδώ και καιρό η ανάγκη μιας πρότασης της Κομισιόν για εναρμόνιση κάποιων πραγμάτων όπως η διάρκεια της αδειοδότησης, ο ορισμός των κριτηρίων αδειοδότησης, επίσης να υπάρχει και για τον κλάδο σαφής κανόνες και αξιοπιστία και ο χρήστης επίσης των κανόνων χρειάζεται κανόνες και πράγματι η εξέταση κάποιων ουσιών ε, απαιτεί πολλές χιλιάδες ευρώ μπορούν να χρηματοδοτηθεί κάτι τέτοιο εάν υπάρχει διασφάλιση ότι δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει και κάποιος άλλος αυτή την ε, ουσία. Πρέπει λοιπόν να προσταμωστούμε και στις νέες απαιτήσει. οπότε θα θέλαμε η Κομισιό να υποβάλει μια σαφή και θεμελιωμένη έκθεση που θα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα ζητήματα κύριε Επιτρόπε και το συντομότερο δυνατόν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο Βιτόριο Πρόντι, ξενόματος των φιλελευθέρων για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, Επίτροπο καταρχήν για την ε, παρουσία του για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό το έγγραφο. Πρόκειται για μία αλλαγή της οδηγίας ως προς τη χρήση βιοκτώνων και το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξουν παρατάσεις επανεξέτασης έτσι ώστε να δούμε τις δραστικές ουσίες ορισμένων βιοκτώνων, λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες αναλύσεις και τις απαιτήσει της αγοράς. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι αναμένουμε μια πιο σοβαρή αναθεώρηση της οδηγίας 98 κάθετος 8 για τα βιοκτώνα έτσι ώστε να έχουμε να κάνουμε με ένα σαφές περιεχόμενο. Θα ήταν σκόπιμο να περάσουμε από μία οδηγία σε ένα κανονισμό, δηλαδή σε ένα κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι δεσμευτικό εξ αρχής για τα κράτη-μέλη, ε, διέποντας ομοιογενώς τον τομέα. Ένα βασικό σημείο είναι το ότι συμμεριζόμαστε και ανταλλάσσουμε τα δεδομένα. Όπως έγινε και με το REACH, έτσι και για τα ε, βιοκτώνα θα πρέπει να μην γίνονται ε, συγκεκριμένες δοκιμές στα σπονδυλωτά και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία από αυτές τις δοκιμές για να μην υπάρχει επικάλυψη στοιχείων. Επίσης, θα έπρεπε να έχουμε μία καλύτερη αξιολόγηση του συστήματος στα πλαίσια της προετοιμασίας για να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της ΜΜΕ και στις εθνικές αρχές που εξετάζουν τις αιτήσει. Θα πρέπει να υπάρχει απλούστευση των διαδικασιών και αμοιβαία αναγνώριση άδειας για το ίδιο προϊόν από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να είναι ταχύτερες οι διαδικασίες ε, χρήσης βιοκτώνων σε διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης θα πρέπει να εναρμονίσουμε και τα τέλη και τον χρόνο εξέτασης των ε, αιτήσεων στα κράτη-μέλη και να απλουστεύσουμε την διαδικασία αδειοδότησης τη στιγμή που υπάρχει μια παρόμοια διατύπωση αποφεύγοντας επιπρόσθετες δοκιμές για περαιτέρω αξιολόγηση από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ Ευρωπαίων παραγωγών με εξοκινοτικούς παραγωγούς. Θα πρέπει η Επιτροπή να εξέβρει μία λύση που να μπορέσει να συμμεριστεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, εξ της Ανεξαρτησίας Δημοκρατίας, η κυρία Κρουπά έχει το λόγο. Η ενοποίηση των, της νομοθεσίας διαβιοκτώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητα ιδιαίτερα καθώς οι κανονισμοί διαφέρουν σημαντικά πράγματα, το οποίο είναι επικίνδυνο και για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε μια φιλελεύθερη αγορά. Το αρχικό έγγραφο με 10 χρόνια περίοδο εφαρμογής δεν είναι ρεαλιστικό λόγο των πολύ δαπανηρών διαδικασιών εγγραφής και αδείας για τα βιοκτώνα. Στόχος είναι βεβαίως η ασφάλεια. Όμως η διαδικασία τελικά υπονομεύει την ασφάλεια διότι σε ορισμένες περιπτώσεις το εθνικό δίκαιο επιτρέπει εγγυήσει για την ασφάλεια παραγνωρίζοντας τους μηχανισμούς και εισαγάγοντας ανεπαρκείς μηχανισμούς και μειώνοντας και το εμπόριο για τα βιοκτώνα. Ε, οι ενεργές ουσίες και ο κατάλογος της κεντρικής Ευρώπης, μάλλον ένας κεντρικός κατάλογος για την Ευρώπη ε, τέτοιων δραστικών ουσιών, ε, δεν θα είναι επαρκής γιατί οι μεταβολές είναι πολύ γρήγορες. Και υπάρχει και μία αντίσταση στην αντικατάσταση. Μικρές εταιρείες μπορεί να εξαφανιστούν τελείως από την αγορά και να δημιουργηθούν και μονοπόλια από μεγάλες επιχειρήσεις. Η μεταβατική περίοδος των 14 συν 2 ετών είναι ουσιαστικότατη ιδιαίτερα καθώς η εγγραφή των ενεργών ουσιών και η μετατροπή του δικαίου του κοινοτικού σε εθνικό δεν είναι εύκολο να γίνει. Πρόεδρος, τώρα έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση για τον Επίτροπο, γιατί έχω μία διαφορετική γνώμη. Λυπάμαι που άκουσα ότι η Κομισιό μας λέει ότι δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εγγραφή των 900 ουσιών βιοκτώνων που, για τα οποία υπάρχει εμπορία στην ευρωπαϊκή αγορά μέχρι το 2010. Μου κάνει εντύπωση που θα χρειαστούμε ακόμη τρία χρόνια. Και η συγγήτρια πρόσθεσε και ένα τέταρτο. Αυτό σημαίνει παράταση ε, στην ανάγκη εναρμόνισης και, ε, της εμπορίας αυτών των ουσιών. Ίσως θα ήταν ε, χρήσιμο κάποιες ουσίες που προέρχονται από την ασιατική αγορά χωρίς να ελέγχονται να ηγηθούν της αγοράς μας και μπορεί επίση να επιταχύνουν την δημιουργία ασφαλιστέρων ουσιών. Ε, θα χρησιμοποιήσει η Κομισιόν τα εργαστήρια των κρατών μελών για να ανταποκριθεί στις προθεσμίες. Θα ήθελα μια απάντηση. Και τώρα ο κύριος Ιστκεύσκη. Λόγω της συγκεκριμένης φύσης και των απειλών που προκύπτουν από την κακή ερμηνεία των νομοθετημάτων για τα βιοκτώνα, τα βιοκτώνα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ο εισηγητής είπε ότι το, η μεταβατική περίοδος μέχρι το 2014 για την εκτίμηση των δραστικών ουσιών που βρίσκονται στα βιοκτώνα είναι απαραίτητη για την τελική ρύθμιση της αγοράς. Οι ε, νόμοι και οι διατάξεις που θα πάψουν να ισχύουν το 2010 μπορεί να οδηγήσουν ε, στην παράνομη χρήση ορισμένων βιοκτώνων κατά τη μεταβατική περίοδο. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχει εθνική εποπτεία της αγοράς κατά αυτή τη μεταβατική περίοδο. Όσον αφορά τα βιοκτώνα λοιπόν, θα πρέπει να λάβουμε προφυλάξεις διότι αυτά τα προϊόντα καταστρέφουν έντομα και άλλους ζώντες οργανισμούς τα αποτελέσματα μπορεί να μην μπορούν να ανατραπούν αν καθυστερήσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, και τώρα πηγαίνουμε ε, στον Επίτροπο, τον κύριο Δήμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές για τις ε, επικοδομητικές τους παρεμβάσεις και θα ήθελα να πω ότι ε, πράγματι η αξιολόγηση των ε, δραστικών ουσιών ε, απαιτεί τελικά περισσότερο χρόνο από ό,τι με αισιοδοξία είχε αρχικά προβλεφθεί. Το 2000 όταν εγκρίθηκε η νομοθεσία δεν άρχισε αμέσως τα προγράμματα αξιολόγησης αλλά περάσανε περίπου τέσσερα χρόνια με διάφορες διαδικασίες προετοιμασίας και μόλις το 2004 ξεκίνησαν οι διαδικασίες ε, ε, αξιολόγησης οι οποίες χρησιμοποιούν αναμφίβολα τις ε, τοπικές, τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Και ενώ έχει γίνει αξιόλογη εργασία και πολύ σημαντική εργασία μέχρι τώρα, εν δεν θα είναι δυνατόν μέχρι το Μάιο του 2010 για πολλές από τις δραστικές ουσίες ε, να έχουν περάσει από την αξιολόγηση. Και δεδομένου ότι η οδηγία ορίζει ότι τα βιοκτώνα προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες μη εγγεγραμμένες στο παράρτημα 1 ή 1α ε, της οδηγίας πρέπει να έχουν αποσυρθεί από την αγορά το αργότερο ως 14 Μαΐου 2010, κρίθηκε αναγκαία να παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης. Διαφορετικά, εάν αποσύρουμε ε, ορισμένες από αυτές τις ουσίες ε, επειδή δεν πέρασαν από τη διαδικασία αξιολόγησης τότε μπορεί ε, να κινδυνεύσει και η υγεία και το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμφίβολα θα υπάρξει και μια παρεμπόδιση του εμπορίου. Για το θέμα το οποίο, στο οποίο αναφέρθη η κυρία Κλάς θα ήθελα να πω ότι το ζήτημα αυτό αφορά την προστασία των δεδομένων που υποβάλλονται για την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας. πρόκειται ειδικότερα για την περίπτωση κατά την οποία εταιρείε οι οποίες δεν έχουν συμβάλει στην προσπάθεια παραγωγής των εν λόγω δεδομένων μπορούν παρά να διατηρήσουν το προϊόν τους στην αγορά μέχρι τη λήξη μεταβατικής περίοδου. είναι οι free riders. η επιτροπή βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας πρότασης ουσιαστικής αναθεώρησης της οδηγίας και πολλές από τις παρατηρήσεις τις οποίες έκαναν οι κύριοι ε, Πρόντι και άλλοι ε, θα ληφθούν υπόψη αναμφίβολα ε, πρόταση ουσιαστικής αναθεώρησης της οδηγίας για τα βιοκτώνα και το ζήτημα αυτό έχει επισημανθεί ξεκάθαρα στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαμόρφωση και διατύπωση σε λόγο πρόταση η επιτροπή θα αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της ουσιαστικής αναθεώρησης οδηγίας. σχετική δήλωση της επιτροπής ε, διαβιβάζεται στη γραμματεία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για καταχώρηση στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίας. επίσης στην εν λόγω πρόταση αναθεώρησης θα αντιμετωπιστούν και πολλά άλλα ζητήματα που έχουν επισημανθεί από το κοινοβούλιο όπως η επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε είδη και υλικά επεξεργασμένα με βιοκτώνα η βελτίωση των διαδικασιών έγκρισης των βιοκτώνων προϊόντων η θέσπιση της υποχρεωτικής ανταλλαγής δεδομένων κατά την αδειοδότηση του προϊόντος και κατά την έγκριση της δραστικής ουσίας σύμφωνα με τις αρχές του κανονισμού reach η ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές άλλων νομοθετικών πράξεων όπως είναι αυτή που θεσπίστηκε πρόσφατα για τα φυτοφάρμακα. καταλήγοντας ε, κύριε πρόεδρε η επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκβαση των διαπραγματεύσεων. η επιτροπή είναι σε θέση να κάνει πλήρως δεκτές τις προτινόμενες συμβιβαστικές τροποποιήσεις και δεσμεύεται να λάβει υπόψη κατά τη διάρκεια της κύριας αναθεώρησης της οδηγίας τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων που εκφράστηκαν ε, τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Κοινοβούλιο και απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Σάρμπου για δύο λεπτά, η συγγήτριά μας για να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο τους κοιόδης επίσης συνεργαστήκαμε αποτελεσματικά και ήμασταν ιδιαίτερα αποδοτικοί στη συγγραφή αυτής της έκθεσης. Βεβαίως η αναθεώρηση της οδηγίας είναι ύψης της σημασίας. Όλοι μίλησαν για αυτή την αναθεώρηση και εγώ για την, έκθεση, την έκθεσή μου, διότι αναμένουμε αυτή την ε, αναθεώρηση της οδηγίας. Ελέγχθη ότι αυτή η παράταση της ε, προθεσμίας κατά τρία έως τέσσερα χρόνια, ε, δεν είναι, από τρία σε τέσσερα χρόνια, ε, δεν είναι επιθυμητή, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα τεθούν στο εμπόριο νομίμως αυτά τα προϊόντα και θα υπάρχει μια σωστή αξιολόγησή τους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και αναμένουμε με αδημονία την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας για τα βιοκτώνα. Λίγη συζήτηση της κοινή συζήτησης και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο.